Κυρίε και κύριοι, γερμανικά και αγγλικά τα λέει ο πρόεδρο. Καθίστε παρακαλώ. Η προετοιμασία αυτής της έκθεσης εμπλέκει επιτροπές όπως και υπό Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας αλλά και την Επιτροπή Προϋπολογισμών και θέλω να καλωσορίσω τον συνάδελφό μου, τον Ζων Αρτουί. Θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το κοινό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, λέει ο κύριος Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Μπροκ. Έχετε κάποια σχόλια από, τους, από την πλευρά, υπάρχουν κάποια σχόλια από την πλευρά των εισηγητών. Κύριε Τάραντ, ούτε και εσείς. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Καλώς. Συμβαστή τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Καλημέρα σας. Συμβαστική 1 υπέρ. The man we're talking about and which is number one on the agenda. Μιλάμε για την έκθεση σε σχέση με τη χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ναι. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ και 27 βέβαια κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά 30 επαναλαμβάνω υπέρ κατά θέλετε έλεγχο καλώς Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 31 με 25 εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Φαντάζομαι θα είναι η ίδια πλειοψηφία. Abstimmung Πέρας. κύριε Φλέκενστάιν. Ε, 30, 33 έχει εκπέσει, 34 ψήφι υπέρ. Την 32 δεν ψηφίσαμε, λέει η γραμματεία. Την ξεχάσαμε. 32 λέει ο πρόεδρος, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μόνο το πρώτο τμήμα λοιπόν έχει εγκριθεί. Σαράντα πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρας. 26 με 42 απερίφθηκε. 27, 27 με 42. 53 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Η άψιμος της... πέρας. 32 32-36 απερίφθη. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές, μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της 71 άρχεται. Πέρας. 32-41 απορρίπτεται πράγματι. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74 σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος. 30 προς 45 απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος Ζητείτε. 77. Έλεγχος. Πέρα της 49 με 22. Εγκρίνεται. Ποιος ήθελε λοιπόν έλεγχο. Ρωτάει ο πρόεδρος. Θα μπορούσα να το φανταστώ λοιπόν. 78. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 80. Υπέρ. Α, εκπίπτει, εκπίπτει, πράγματι. Πάμε στην 82. Υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 και 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ τελικά. Την 106 την ψηφίσαμε, πράγματι. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 και 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 117 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται 118 υπέρ με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1.21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 122 υπέρ. Πώς είπατε? 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Εγκρίνεται. Η επτά εκπίπτη υπέρ κατά αποχές. Οκτώ υπέρ έλεγχος για την οκτώ. Πέρας πληροφορίας. 32-43 απορρίπτεται. Εννέα. Ή οχτώ. Απερίφθη λοιπόν. <clears throat> Εννέα. Κατά αποχές συγκρίνεται. Δέκα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή, Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και ερχόμαστε τώρα στο σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. 54 εναντί 23 με δύο αποχές γίνεται δεκτή. Δεν γίνεται δεκτό το ψήφισμα. Κύριε Κόουζο, απλώς θα να σας πω ότι η ΓΚΟΕ NGL ψήφισε κατά γιατί δεν συμμεριζόμαστε τη γενική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει μια έκθεση μειοψηφίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δικαίωμα ασφαλώς να την υποβάλλατε. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Θα να χαιρετήσω την εργασία των ε, συνεισηγητών και πραγματικά να χαιρετήσω και την ποιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μας επιτροπές. Thank you.